ψηφίσματα, αλλά θα αρχίσουμε με την Επιτροπή. Παρακαλώ, Ο Επίτροπος Έτσιγκερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί το Κοινοβούλιο για τη δυνατότητα που δίνει να διεξαχθεί η συζήτηση αυτή να συζητηθεί η Σρεμπρένιτσα με την ευκαιρία αυτού ψηφίσματος που έχετε καταθέσει. Πρόκειται για μια σημαντική κοινή δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων 20 χρόνια μετά τα φρικτά αυτά γεγονότα μπορούμε να μνημονεύσουμε τα θύματα και να σταθούμε στο πλευρό των οικογενειών και των οικείων τους που έχασαν τους αγαπημένους τους. Και πρέπει να φροντίσουμε εφ' να γίνεται οτιδήποτε είναι δυνατόν για να προστατεύονται τα θύματα. Η γενοκτονία της Ρεμπρενίτσα έχει στιγματίσει όχι μόνο την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και για μας όλους επιβάλλει τη διαρκή ηθική ευθύνη να μην λησμονήσουμε. Απαιτεί από όλους μας και ιδιαίτερα από τους ερετούς ε, πολιτικούς και εκλεγμένους προσώπους της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης και ολόκληρης περιοχής να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προσταθούν στη δικαιοσύνη οι υπέτη των εγκλημάτων πολέμου αλλά και να πραγματοποιηθούν ουσιαστικά βήματα συμφιλίωσης σε ολόκληρη την περιοχή για το καλό της τωρινής και των μελλοντικών γενναίων. για να απαλυνθεί ο πόνος των οικείων των θυμάτων, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπέτοι και να βρεθούν οι ακόμα αγνοούμενοι. Πρόκειται για εκ όρο για μια μακροπρόθεσμη και διαρκή συμφιλίωση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και ολόκληρη την περιοχή μεταξύ των διαφορών λαών που ζουν εκεί. για τους ε, υπεύθυνου εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η Σρεμπρένιτσα ήταν ένα μάθημα ότι δεν θα πρέπει να αφήνουμε στη μοίρα τους περιοχές τέτοιες και γι' αυτό βλέπουμε τώρα τα Δυτικά Βαλκάνια υποψήφια ε, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, με μια διαδικασία αξιόπιστων μεταρρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων αποκατάσταση εμπιστοσύνη των πολιτών μεταξύ τους, στη Βοσνία αλλά και την ολο... γενικότερη περιοχή. Και εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι η μνήμη της Ρεμπρέντσα πρέπει πάνω απ' όλα να τιμά τα θύματα της ε, γενοκτονίας αλλά ταυτόχρονα να ανοίγει το δρόμο για τη συμφιλίωση στη Βοσνία αλλά και σε όλα τα κράτη της περιοχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει να προχωρήσουν οι πολιτικοί και οι κοινωνίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο καλύτερος δρόμος για να μπορέσουν να αφήσουν πίσω τους τα εγκλήματα και την τραγωδία αυτή. Όχι να τα ξεχάσουν, να τα αφήσουν πίσω τους. Και να μην επανληφθούν τέτοιου είδους εγκλήματα και τραγωδίες. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σημερινό του ψήφισμα και εκφράζεται τη λύπη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ένα αντίστοιχο ψήφισμα που κατατέθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετώπισε το, την έγερση αρνησικυρίας εκ μέρους της Ρωσίας δυστυχώς και έτσι δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Τέτοιου είδους πράξεις δεν μπορούν να ε, αξιοποιούνται πολιτικά εις βάρος της μνήμης και εις βάρος της συμφιλίωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πρέντα έχει τώρα το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Το ψήφισμα, το κείμενο που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως σε ένα πλαίσιο από το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών χτες δεν μπόρεσε να εγκρίνει ψήφισμα οφείλουμε να τιμήσουμε τα θύματα αυτών των απεχθών εγκλημάτων που έλαβαν χώρα 20 χρόνια τώρα στη Σρεμπένιτσα. Η σκέψη μας λοιπόν σήμερα πάει στα θύματα και στις οικογένειές τους. Είναι χρέος μας, χρέος μνήμης, εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Χωρίς αυτό το έργο μνήμης δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση εξάλλου αν δεν μάθουμε την αλήθεια όσο και αν αυτή πονάει. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ και 20 χρόνια έλαβε χώρα μια γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και εμείς την καταδικάζουμε. Και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται να ελαφρύνουμε τα βάρη, γιατί αυτό πλήττει και τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και τη διαδικασία συμφιλίωσης. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους πολιτικούς ηγέτες στην Βοσνία Ριζεγοβίνη και σε ολόκληρη την περιοχή προκειμένου να αποτελέσουν παράδειγμα, να αναγνωρίσουν αυτό το δύσκολο παρελθόν προκειμένου η χώρα τους να μπορέσει να πάει μπροστά. Εμείς από τα δικιά μας την πλευρά πρέπει να φροντίσουμε να μην ξανά έχουμε τέτοια γεγονότα. Να στηρίξουμε την ακερότητα την ολοκλήρωση τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και των Βαλκανίων και είναι ο καλύτερο τρόπο για να του βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν του διχασμού του. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φαγιών έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, Θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι νομίζω αλληλέγγυοι μέσα σε αίσθημα σεβασμού των ανθρώπων. Παρακαλώ συνεχίστε. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Μπορείτε όμως τώρα να συνεχίσετε. Πριν από 20 χρόνια η Ευρώπη σφάδαζε από τους ε, πολέμους σε ένα μέρος της ε, Ευρώπης λοιπόν ε, έχουμε όμως τώρα δει ότι μπόρεσε να προχωρήσει και το κράτος δικαίου και η δημοκρατία και η ειρήνη η συμφιλίωση είναι ο σημαντικότερο στόχο. Ε, φυσικά η μνήμη είναι πολύ σκληρή. 8.000 Βόσνοι έχασαν τη ζωή του στη Σρεμπρένιτσα πριν από 20 χρόνια. Και πρέπει να βρούμε μία λύση για τη συμφιλίωση. Ο Σρέντερ την 60η επέτειο του Auschwitz είπε ότι πολλοί θέλουν να λησμονήσουμε αλλά δεν πρέπει να λησμονήσουμε. Το ίδιο ισχύει και στην Σρεμπρένιτσα. Δεν θα λησμονήσουμε τα θύματα της γενοκτονίας εκεί αλλά και οπουδήποτε αλλού στη Ιουκοσλαβία. Γιατί δεν θα υπάρξει ούτε ελευθερία, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε ειρήνη αν λησμονήσουμε τα θύματα ή κλείσουμε τα μάτια μας. Η Σρεμπρένιτσα πρέπει να εξακολουθεί να μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ακόμα μένουν πάνω από χίλια αγνοούμενοι. Αυτούς θα τους θυμίσουμε το επόμενο Σάββατο και εγώ θα ήθελα σήμερα να καλωσορίσω το ψηφισμά που έχουμε να εγκρίνουμε. Η περιφερειακή συνεργασία και η προσέγγιση της Βοσνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσει το διχασμό και το μίσος. Λυπούμε που δεν μπόρεσε το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών να υιοθετήσει το ψήφισμα για τη Σρεμπρένιτσα. Νομίζω ότι θα πρέπει σε, ενώπιον τέτοιων ζητημάτων να ξεπερνάμε τα πολιτικά συμφέροντα και τους φραγμούς. Πρόκειται για ηθική υποχρέωση ηθική υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε την Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Τόματσις. Η κυρία Τόματσις. Ευχαριστώ. Αυτή την εβδομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο ε, θυμόμαστε το γενοκτονία στη Σρεμπρενίτσα, εστιαζόμαθα στα θύματα και τα όσα πέρασαν οι οικογένειές τους. Αλλά δράτω με αυτή τη θλιβερής επαιτίου για να υπενθυμίσουμε, υπενθυμίσουμε σε αυτούς μας το θλιβερό ρόλο που διαδραμάτισε η διεθνής κοινότητα σε αυτή την φρικτή αιματοχυσία. Ε, σχεδόν τέσσερα χρόνια πέρασαν μεταξύ Μπούκοβαρ και Σρεμπρενίτσα Δυστυχώς όμως αυτή η χρονική περίοδος δεν ήταν αρκετή. Καταστράφηκε ολοσχερός το Μπούκοβαρ. Δολοφονήθηκαν άμαχοι και υπήρχαν στρατόπεδα για Κροάτες στο έδαφος της Σερβίας. Όλα αυτά όμως που ήταν γνωστά δεν άνοιξαν τα μάτια του κόσμου για να καταλάβει τις βιοπραγίες που λάμβαναν χώρα στην Κροατία. Τα αποτελέσματα ήταν τα χειρότερα δυνατά μερικά χρόνια αργότερα. Είχαμε τη Σερμπρενίτσα. Και όλοι αυτοί που θέλουν να σχετικοποιήσουν τα πράγματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μόνο η αλήθεια οδηγεί στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη στην εσωτερική γαλίνα. Γαλήνη, συγγνώμη. Βέκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριος Γιάκοβιτς. Εδώ και 20 χρόνια στην Σερμπρένιτσα, διπράχθη γενοκτονία τα πιο φρικτά εγκλήματα πολέμου μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε έδαφος ευρωπαϊκό. Τα κίνητα του εγκλήματος ποια ήταν, ότι απλώς ο άλλος ανήκε σε κάποια άλλη θρησκεία ή άλλη εθνικότητα. Και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, διότι ζούμε βάσει κοινών αξιών που μας ενώνουν. Και οι πολιτικοί στη Βοσνία Ζεγοβίνη αυτό θα πρέπει να το παραδεχθούν. Ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η διχόνοια στη Βοσνία Ζεγοβίνη και ήρθε η ώρα να δεχτούν ότι η Ευρώπη του στέλνει ε, μαζί τη. Και ήρθε η ώρα να ποτίσουμε φόρο τιμή εκείνου στη Βοσνία Ζεγοβίνη στα θύματα και σε όλες εκείνες τις οικογένειες που ακόμα υποφέρουν σήμερα. Όλες οι πλευρές στη Βοσνία εζεγοβινη διέπραξαν φρικτά εγκλήματα. Δυστυχώς και μέλη της δικής μου χώρας και θα πρέπει να είμαστε αρκετοί γενναίοι να πούμε ποια είναι η αλήθεια, να δεχτούμε την αλήθεια. Η Σρεμπρένιτσα εξακολουθεί να είναι σύμβολο τραγωδίας και θλίψης για όλο το λαό της Βοσνίας εζεγοβινης και γι' αυτό αυτή η μέρα θα πρέπει και στο μέλλον να είναι επέτειος θα πρέπει να είναι μια επέτειος που θα αποτείουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που υπέφεραν εκεί στην, στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, ο καθένας από εμά θα πρέπει να διερωτηθεί. Θα πρέπει να δει κατά πόσο θα μπορούσε να έχει σταματήσει τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι η διεθνής ε, κοινότητα απέτυχε παταγωδός να κάνει αυτά που προσδοκούσαν σε όλο τον κόσμο και να αποφευθεί η σφαγή της Ρεμπρένιτσα. Οι ένοχοι θα πρέπει να τιμωρηθούν και περιμένω το δικαστήριο της Χάγης να εκτελέσει το καθήκον του. Λυπούμε διότι ο ΙΕ δεν είχε το θάρρος να εθετήσει ψήφισμα διότι το περιμέναμε όλοι αλλά είναι καλό ότι εμείς έχουμε εδώ κοινό ψήφισμα. Ε, και κάτι άλλο που είναι καλό δηλαδή η απόφαση να μεταβούμε στη Σρεμπρενίτσα. Αυτό δεν είναι ένα ψήφισμα που είναι κατά τη Σερβία ή κατά των Σέρβων. Είναι ένα ψήφισμα που προσπαθεί να βοηθήσει τη Σερβία να αντιμετωπίσει την αλήθεια και στο τέλο όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ράνστοφ. Κύριε Ράνστοφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε συμβεί ποτέ εάν οι Αμερικανοί δεν είχαν βάλει τον Ιζαμπέκοβιτς να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρθηκε απέναντι στις συμφωνίες του 1992. Το δεύτερο τώρα για τον Κάρατσιτς. Δεν μιλάμε για αυτόν που τα έκανε όλα αυτά που είναι ο Νάσερ Ρόριτς, ένας επιχειρηματίας από την Τούσλα, ο οποίος το 2006 ελευθερώθηκε στη Χάγη. Γιατί όλοι οι μάρτυρες είχαν εξαφανιστεί, ήταν αγνοούμενοι ή είχαν σκοτωθεί. Και επειδή δεν υπήρχαν λοιπόν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, ελευθερώθηκε στη Χάγη. Φυσικά πρέπει να τιμούμε τη μνήμη, αλλά δεν είναι το τέλος αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Σόλτες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να θυμηθώ βέβαια όλους όσοι δολοφονήθηκαν στη Στρεμπέντσα. Αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αλήθεια. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλοι. Και μια μεγάλη ευθύνη είναι και στους διεθνείς οργανισμούς. Τα δικαστήρια πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους βέβαια. Και εμείς τιμούμε τα θύματα. Τις μανάδες που είδαν τους γιους τους, τους άντρες τους, τους αδερφούς τους να δολοφονούνται. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξεπεράσουν τις προσπάθειες που γίνονται για να ξεχαστούν όλα αυτά. Πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη για τις οικογένειες αυτές. Όπως επίσης και για εκείνους το όνομα των οποίων έγιναν οι σφαγές και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη σφαγή. Γιατί και αυτοί πρέπει να μπορέσουν να γυρίσουν σελίδα και να ζήσουν μέσα σε μια πολυεθνική κοινωνία. Προκειμένου η Βοσνία να μπορέσει να νίκει εκεί που πραγματικά νίκει, δηλαδή στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Συνοδεινός έχει το λόγο. Μνήμης όπως αυτή της Ρεμπρέντζα έχουν σαν σκοπό να θυμίζουν και να διδάσκουν στις νεότερες γενιές το έβρος της ανθρώπινης θηριωδίας που τρέφεται κυρίως από τον εξτρεμισμό. Να παραδειγματίζουν και να λειτουργούν αποτρεπτικά. Δυστυχώς όμως τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα διαπράττονται σήμερα από τους συγχαντιστές δολοφόνους Αλκάιντα, της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού κράτους η σρεμπρένιτσα όμω δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονό. ήταν αποτέλεσμα τη ομή παρέμβαση των αμερικανών και γερμανών που επιθυμούσαν τη διάλυση της ενωμένης για γεωπολιτικού ιδιωτελεί σκοπού. ήταν εγκληματική επίθεση εναντίον ενό κυρίαρχου κράτου που αποτελούνταν από σλαβικέ εθνότητε. τα άσχημα αποτελέσματα τη πολιτική αυτή τα βλέπουμε μέχρι σήμερα. τη βοσνία ερζεγοβίνη των τριών διαφορετικών εθνοτήτων που μισεί η μία την άλλη; το κωσυφοπαίδιο όπου υπήρξε βίαιο εκτοπισμό των σέρβων και παράνομο επικισμό από αλβανού τη φύρομ ένα κράτο συνοθήλευμα εθνοτήτων με ονειρόξει κλοπή του ελληνικότατου ονόματο μακεδονία. οι μέρε μνήμη είναι ιστορία. την ιστορία δεν πρέπει να την παραγράφουμε ούτε να την παραποιούμε. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πλέκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα τιμούμε τα 20 χρόνια από τη σφαγή της Ριμπρένιτσα. Και θέλω εδώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τις οικογένειες των θυμάτων. Εμείς καταδικάζουμε την γενοκτονία αυτή που έγινε από τις σερβικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Ράτκον Πλάντιτς. Το 1995, όταν πάνω από 8.000 αγόρια και άντρες μουσουλμάνοι δολοφονήθηκαν. Το 1997 είπαμε ότι η Σερβία δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει τη γενοκτονία αυτή. Ελπίζουμε λοιπόν το δικαστήριο της Χάγης να δράσει. Χτες η Ρωσία δεν ψήφισε το ψήφισμα και υπήρχαν και αποχές, Βενεζουέλα, Κίνα. Το ψήφισμά μας λοιπόν πρέπει να προχωρήσει και να μην σχετικοποιούμε τα γεγονότα, να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει εκεί. Πιστεύω ότι η συμφιλίωση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον ξέρουμε την αλήθεια, την παραδεχτούμε και μόνο αν συγχωρήσουν τα θύματα. Διότι χωρίς αμφιβολία Όλα αυτά παρέουν από τον Μιλόσεβιτς και όχι μόνο στη Βοσνία Ζηγοβίνη. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Σκάνης. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την εβδομάδα έχουμε την επέτειο, την 20η επέτειο από τη γενοκτονία της Ρεμπερενίτσα. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και αποτείμε φόρτι στους, στους, ε, στις 42 οικογένειες που ζητούν δικαιοσύνη. Είναι ντροπή για τον κόσμο. Δεν μπόρεσε να προστατεύσει αθώους ε, άμαχους πολίτες. Κυρία Πρόεδρε, είναι απογοητευτικό που ο ΙΕ δεν πέρασε το ψήφισμα, κυρίως όταν το Διεθνές Δικαστήριο είχε ε, αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Θα πρέπει να μαθαίνουμε το παρελθόν, ανανεώνουμε την αποφασιστικότητά μας, ποτέ να μην αφήσουμε την προκατάληψη, το μίσος και το κακό να δρουν ανενόχλητα. Θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά κρατούμε τα μάτια μας ε, προς το μέλλον της Βοσνίας. Η συμφιλίωση παραμένει θεμελιώδης στόχος. Αυτό το μονοπάτι περνάει μέσα από τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Η συμφιλίωση παραμένει θεμελιώδης στόχος και αυτό το μονοπάτι οδηγεί στη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Θα πρέπει να προωθήσουμε την εκπαίδευση, την ανάμνηση και την έρευνα για τα γεγονότα αυτά στη Σρεμπρενίτσα και για άλλες γενοκτονίες. Οι μελλοντικέ γενιές θα πρέπει να καταλάβουν ποια είναι τα αίτια τέτοιων σφαγών και θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινωνίες που βασίζονται στην ένταξη, στην αλήθεια και θα πρέπει η Βοσνία Ζεγοβίνη να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Το ευρωπαϊκό μονοπάτι είναι ο καλύτερο τρόπο να προχωρήσει κανεί πέρα από τι τραγωδίε του παρελθόντο. Παροτείνουν οι ηγέτε να συνεργαστούν ούτω ώστε η χώρα να γίνει ασφαλή και να επικρατήσει ευημερία. Γι' αυτό θα αποτείουμε φόρο τιμής στα θύματα της Εμπενίτσα. Πάντα η σκέψη μας και η καρδιά μας ε, θα στρέφεται προς αυτούς. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Λούνατσέκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Σάββατο εκ μέρου του Προέδρου Σούλτ θα εκπροσωπήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με 10.000 άλλου που θα πάμε στη Σρεμπρένιτσα για τι ε, εκδηλώσει μνήμη. Θα μεταφέρω τις εκδηλώσεις τιμής και σεβασμού προς τα θύματα και τα συλληπιτήρια προς τους επιζήσαντες. Θα τα μεταφέρω μαζί μου από εσά εδώ. Ύστερα από το αποτροπιαστικό αυτό έγκλημα μπορώ να πω ότι χαίρομαι που μπόρεσε το Κοινοβούλιο να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων και λυπούμε που στα, που στα Έθνη ε, υπήρξε παρεμπόδιση του ψηφίσματος. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμη το δικό μας ψήφισμα. Η ειρήνη μπορεί να απέλθει μόνο όταν μιλούμε για την ε, φρικαλαιότητα, όταν καταδικάζουμε τα εγκλήματα, όταν μπορούμε να προχωρήσουμε και προς τη μνήμη βέβαια και προς τη συμφιλίωση όμως. Θα ήθελα επίσης να τιμήσω τις γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού και των οποίων τα δεινά και ο πόνος δεν έχουν αναγνωριστεί παντού. Δεν πρέπει ποτέ να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Στην Ήπειρό μας ή σε οποιαδήποτε άλλη Ήπειρο δεν πρέπει ποτέ να συμβούν αυτά που συνέβησαν στη Σρεμπρίνιτσα. Ευχαριστώ πολύ, Πίκουλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Περιμένουμε ίσως ε, να πάρουμε αποστάσεις χρονικές από τα ιστορικά γεγονότα για να μπορέσουμε να δούμε πιο καθαρή εικόνα. Αυτό που συνέβη όμως στην Ρεμπρένιτσα ήταν γενοκτονία και δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Μια σειρά από τραγωδίες του 20ου αιώνα ξεκινάει από μια πόλη πολύ κοντά στη Ρεμπρένιτσα, το Σαράγεβο. Ξεκίνησε με το πρώτο, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος από το Σαράγεβο, όπως και τέλειωσε το 1995 στη Σρεμπρένιτσα. Αυτό που καθιστά ακόμη πιο τραγική τη μοίρα των ανθρώπων αυτών είναι το γεγονός ότι αντίθετα από ό,τι συνέβαινε στι αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε ένα συλλογικό σύστημα εθνών το οποίο θα έπρεπε να μπορέσει να αποτρέψει την ε, ασυγκράτητη βία και μίσος που έφερε τόσα θύματα. Τώρα 20 χρόνια μετά προσπαθούν μέσω της ε, σιωπή και του κινησμού ορισμένοι να ξανασκοτώσουν τα θύματα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αισθάνεται υπερήφανο για την συμβολή του και το ψήφισμα το οποίο θα εγκρίνουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή πριν από τη διαδικασία ο κύριο Κρέλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενωμένοι στην ε, διαφορετικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να φτάσει και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για το καλό των πολιτών εκεί, για το καλό των νέων εκεί, για την ειρήνη, για την περιοχή και για το μέλλον όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πριν από 20 χρόνια έλαβε χώρα ένα από τα χειρότερα εγκλήματα εκεί. Η γενοκτονία, ο εθνικός ε, για την κάθαρση. Χιλιάδε ήταν οι αγνούμενοι στη Σεμπρέβιτσα, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στην Κροατία. Για το καλό λοιπόν των μελλοντικών γενεών πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειές μα προκειμένου να μπορέσουν να συμφιλωθούν όλοι στην περιοχή και να έχουν ένα μέλλον. Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλου του θεσμού και σε όλου του πολίτε τη Βοσνία Ερζεγοβίνης να διπλασιάσουν τι προσπάθειές του προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο. Κύριος Κούκαν είναι ο πρώτος. Παρακαλώ κύριε Κούκαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με Δέος θυμούμε τη μνήμη αυτών, αυτών που έχασαν τη ζωή τους πριν από 20 χρόνια. Εκφράζουμε τη λύπη μας στους οικείους τους και τα συλληπιτήριά μας. Ο πόνος των ανθρώπων εκεί είναι δικός μας πόνος και δεν πρέπει κανείς να λησμονήσει τη γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα. Ηθικό μας καθήκον είναι να εξακολουθούμε να τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων αυτών και να λέμε ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δε όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα φορούν στο πέτο το λουλούδι της Τρεμπρένιτσα, το άνθος της Τρεμπρένιτσα, σαν σύμβολο μνήμης. Και πρέπει νομίζω να αποτελέσει αυτό μια ευκαιρία να αναστήσουμε τη συμφιλίωση στη ε, Σρεμπρένιτσα και τη Βοσνία Σεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα θυμόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτά που συνέβησαν στη Βοσνία Ζεγοβίνη, τους ανθρώπους εκείνους που δολοφονήθηκαν. Δυστυχώς, τα στατεύματα του ΟΗΕ δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τον κόσμο. Ενώ αυτό ήταν το βασικό τους καθήκον θα πρέπει αυτό να το ελέγξουμε με τον ΟΗΕ, με τις συνευτικές δυνάμεις. και τις συνευτικές δραστηριότητε. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Αυτό να μην ξανασυμβεί. Πρέπει να καταγγείλουμε ότι καταψηφίστηκε το ψήφισμα στον ΟΗΕ για το γενοκτονία πλευράς Ρωσίας. Είναι απίστευτο. Πώς μια χώρα μπορεί να αρνηθεί αυτή τη γενοκτονία. Οι ένοχοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Η συμφιλίωση είναι σημαντικότατη για τη Βοσνία Ζεγοβίνη στο δρόμο της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτού του είδους η γενοκτονία δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, στην 20η επέτειο τη σφαγή Σρεμπρενίτσα είναι σημαντικό αυτή η γενοκτονία που διεπράχθη κατά 8.000 Βοσνίων μουσουλμάνων, ανδρών και παιδιών και ανδρών και αγοριών να τη θυμόμαστε στη χειρότερη φρικαλαιότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Χίλια αγόρια και άντρε είναι ε, αγνοούμενοι και υποτίθεται ότι έχουν ε, θαυτεί αφού έχουν εκτελεστεί εμψυχρό από τις ε, βοσνιακές σερβικές δυνάμεις και ο ΙΕ αμέλησε την, ε, το καθήκον του να προστατεύσει τους αμάχους στην περιοχή και θα ήθελα όπω και άλλοι συνάδελφοι να πω ότι συγκλονίστηκα από την ανησυχία τη Ρωσία, κατά τη βρετανική κυβερνήση που προσπάθησε να περάσει ένα ψήφισμα τη Αμπερνίτης από το Συμβούλιο Ασφαλεία στο ΙΕ. Τα αγωδίε αυτού του είδου ποτέ δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικού ποδοσφαίρου. Η Ρωσία δεν έμαθε τα μαθήματά τη από τι σφαγέ στο Κατίν κατά τη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είπε ψέματα ο Στάλιν και κατηγόρησε του Γερμανού. Ούτε αυτό θα έπρεπε ποτέ να ξανασυμβεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Συνάδελφε Τσούτσουκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, οι φρικαλαιότητες που έλαβαν χώρα πριν από 20 χρόνια στη Στρεμπρένιτσα μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Όλοι όμως καταλήγουν στο ότι η μετάβαση από τον ολοκληρωτισμό σε δημοκρατικές ε, δημοκρατίες στα Βαλκάνια έχει περάσει από ε, ματοχυσία. Εμείς τα καταφέραμε να κάνουμε τη μετάβαση αυτή χωρίς αιματοχυσία. Είναι το πιο βασικό, πιστεύω, και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Κάναμε ε, να βγουν λάθος οι αναλυτές που έλεγαν ότι στη Βουλγαρία θα καταλήξουμε σε έναν ε, ενδοεθνικό πόλεμο. Δεν έγινε όμως διότι ήταν ξεκάθαρο για μας πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση στα Βαλκάνια. Η τραγωδία λοιπόν στην Ρεμπνεύνητσα είναι για να μας θυμίζει ότι έχουμε ηθικό χρέος απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι εταίροι μας και στηρίζουν την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει Πρόεδρος, Πίντο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το μέγεθος της καταστροφής πριν από 20 χρόνια στη Σεμπρενίτσα μας υποχρεώνει σήμερα να δείξουμε θάρρος και να πούμε ότι οι αθώοι δεν υπάρχουν. Οι μόνοι αθώοι ήταν τα θύματα και οι οικοί τους. Και όπως συχνά συμβαίνει σε τις καταστάσεις, η διεθνής κοινότητα άρχισε να εξασφαλίσει την συμφιλίωση και να ανοίξει το δρόμο για τη συμφιλίωση. Τώρα πρέπει να φροντίσουμε να μην μείνουν ατιμόρυτοι οι υπέτειοι αυτών των σφαγών. πρέπει να τους επιβάλλουμε τις συνέπειες των εγκλημάτων τους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η διεθνής κοινότητα να τιμωρήσει τους υπέτειους των εγκλημάτων. Και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να ε, αναπαυθούν εν ειρήνη οι νεκροί. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Έτιγκερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή συζήτηση είναι, νομίζω, δείγμα της ε, περίφραστης δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της προσήλωσής του στην ειρήνη, στη συμφιλίωση, στη μνήμη της γενοκτονίας Τρεμπρένιτσα πριν από 20 χρόνια. Με την συμμετοχή σας και τη συζήτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δηλώνουν από κοινού ότι τιμούν τα θύματα των σφαγών στη Βοσνία, Ερσεγοβίνη και όλη την περιοχή πριν από 20 χρόνια. Τα γεγονότα αυτά μας υπενθυμίζουν γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα ήταν ένα εγχείρημα για την ειρήνη. Ένα σχέδιο να σταματήσει η διχοτόμηση της Ευρώπης όπως έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα εγχείρημα για να πέσει το τείχος του Βερολίνου ένα εγχείρημα για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζουν σε μια ενιαία Ήπειρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά και βέβαια να ζουν όλοι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο ειρηνικό. Η Βοσνία Σεγοβίνη έχει μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική, της το έχουμε πει. Το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο πολλές φορές δεν θα αφήσουμε οιασδήποτε προσπάθειες για να βοηθήσουμε τα μέλη, τα, τα κράτη το, της περιοχής των Βαλκανίων να ε, προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Έχω 7 αιτήσει για προτάσεις ψηφισμάτων για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Περατώνεται η συζήτηση και θα ψηφίσουν